2 Ιανουαρίου. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες μετά από αυτήν την ανακοίνωση. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο ψήφισμα για τους Ιταλούς, Εσθονούς και Βρετανούς ε, ναυτικούς που ε, κρατούνται στην Ινδία. Έχουμε ε, τις στροπολέξη των πρασίνων. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Αυτό ε, ε, τώρα το, το ENF υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σχέδιο κοινού ψηφίσματος. Ψηφίζουμε το κείμενο συνολικά. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψήσουμε για την Αιθιοπία. Κοινό σχέδιο ψηφίσματος τροπολογίας Γκουε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτω τροπολογία της ΓΚΟΕ. Να ελέγξουμε. Σπραβδάμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται τροπολογία. Τώρα ψηφίζουμε το κείμενο ε, του κοινού το υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, teraz ψήφισμα για τη Βόρεια Κορέα κοινό ψήφισμα αρχικό κείμενο παράγραφος 4 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση, <clears throat> άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Πέρας. Εγκρίνεται. Έχουμε εξαντλήσει τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και σας ε, εύχομαι καλή επιστροφή στις αιστείες σας στα πρακτικά της συνεδρίασής μας. Θα παρουσιαστούν στην αρχή της επόμενης Συνόδου Ολομέλειας και θα θεωρθούν εγκεκριμένα εάν δεν υπάρξει αντίληση. Και τα ψηφίσματα που εγκριθήκαν σήμερα